Ε, η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ε, είπα τη εκπροσώπου τη Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, εν των συνόδων του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών 2016. Η κυρία Μογκερίνη και πάλι έχει τον λόγο παρά. Όπω ξέρετε Πρόεδρε, ταξίδευσα πολύ στον κόσμο κατά τη διάρκεια της μου μέχρι τώρα και είδα την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα μάτια των φίλων και εταίρων. Και όταν μας βλέπουν, σκέφτονται αμέσως δύο πράγματα. Την οικονομική μας ισχύ, ακόμα και μετά την κρίση, ελπίζοντας ότι η κρίση θα έχει περάσει, και τη δουλειά που κάνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm. Θεωρώ την συζήτηση αυτή σαν δυνατότητα να καθορίσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ για το 2016 και πώς θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο και τι σημαίνουν για μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα βασικά εργαλεία είναι να υποστηρίξουν ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Θέλουμε να έχουμε πολυμερή προσέγγιση και επαφέ με όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Γι' αυτό το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κεντρική σημασία. Είναι ένας τομέας όπου μπορεί να ληφθούν αποφάσεις σημαντικές κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι κεντρικός τόπος στον ΟΗΕ για να δημιουργούνται εταιρικέ σχέσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Θέλουμε να προωθήσουμε δικαιοσύνη, ισότιμία, συνεργάσιμες ε, προσεγγίσεις κατά των βιοπραγιών, της καταστολής κλπ. Λοιπόν, θα, θα δώσουμε προτεραιότητε λοιπόν στο Συμβούλιο αυτό τι δύο χειρότερες περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, στην Βόρεια Κορέα θα το συζητήσουμε αύριο ε, στο ημικύκλιο και την Συρία που συζητήσαμε χθε. Λοιπόν, είναι ίσω το πιο καταπιεστικό κράτος ε, στον κόσμο η Βόρεια Κορέα. Ελευθερία έκφραση, θρησκεία και κίνηση, μετακίνηση είναι ανύπαρκτα. Εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι παραμένουν κρατούμενοι σε στατόπεδα πολιτικών κρατουμένων και σε άλλα σημεία που κρατούνται κρατούμενοι. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί από για κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο έγκλημα. Λοιπόν, στο Συμβούλιο αυτό θα συνεργαστούμε με την Ιαπωνία για να ετοιμάσουμε ψήφισμα ε, που θα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Το ψήφισμα θα ζητά ε, λογοδοσία και θα επεκταθεί και η εντολή που θα δοθεί στον ειδικό εισηγητή. Θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην διαδικασία αναθεώρησης που θα εφαρμοστεί για τη Βόρεια Κορέα και για να ξαναξεκινήσει η υποβολή ε, εκθέσεων σε τη μειονότητες στους αρμόδιους φορείς. Η Συρία μετά είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο. Δεν υπάρχει παραλληλισμός στην ιστορία. Πρώτη προτεραιότητα στις συνομιλίες της παρούσες είναι να επιτρέψουμε ανθρωπιστική πρόσβαση στα περισσότερα σημεία της χώρας, στα μεγαλύτερα σημεία της χώρας. Αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στο σχετικό ψήφισμα της Συρία. Η πρόσβαση ε, βοήθειας απεστάλλει στη Μετάγια ήταν ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί από πολλά άλλα βήματα. Μακροπρόθεσμα, η ειρήνη στη Συρία απαιτεί δικαιοσύνη και λογοδοσία για όλους θα πρέπει να συναρμολογήσουμε τα κομμάτια της συριακής κοινωνίας, δεν είναι εύκολο η συμφιλίωση απαιτεί καταρχάς αναγνώριση των δεινών που έχουν περάσει οι Σύριοι και γι' αυτό θα υποστηρίξουμε περαιτέρω επέκταση της εντολής που θα δοθεί στον αρμόδιο, στην Επιτροπή της ε, ε, εξεταστική, διότι είναι το μόνο εργαλείο που συλλέγει στοιχεία για υποστήριξη μελλοντικών μηχανισμών δικαιοδοτικών, δικών. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκεί μπορεί να προωθήσει διάφορες θετικές εξελίξεις. Λοιπόν, μετά θα έχουμε Μιανμάρ, Βυρμανία, όπου εκεί έγιναν ιστορικές εκλογές, οι ιστορικές κρίσεις του Νοεμβρίου είναι βήμα πρόοδου. Έχουμε τη Μογγολία, μετά όσον αφορά εθνοτικές και συσκευτικές μειονότητες, μετά θα παρουσιάσουμε και ένα ψήφισμα όσον αφορά σχόλια για τη νέα κυβέρνηση που αναλαμβάνει καθήκοντα τον Απρίλιο, θα πρέπει να κινηθεί ταχαίως και τολμηρός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και έτσι θα πρέπει να συνεχίζεται έλεγχος ο πλευράς ΟΗΕ των εξελίξεων στη χώρα. Θα παρουσιάσουμε επίσης δύο θεματικά ψηφίσματα, ένα για την ελευθερία της θρησκείας και τον πιστεύω θέλουμε να στηρίξουμε την καταπολέμηση της θρησκευτική μυσαλλοδαξίας υπό ενδήποτε μορφή και έκφραση και μετά θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε προ λίγων ωρών και κοινό τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και Σετική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Παιδιών Ελευθερία ή την Ανεξιθρησκεία θα διοργανώσουμε και κάποια εκδήλωση όπου ειδικό ε, εισηγητής θα παρουσιάσει τα απορίσματα του τα βασικά μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας Συρίας. Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπετε, ε, χωρίς την, ε, μάλλον την παρουσία της κοινωνίας των πολιτών. Όλο το έτος θα συνεργαζόμαστε με τέρους για να προωθούμε και να προωθούμε ε, την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να πω και τον ρόλο των πρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διαδικασίες του ΟΗΕ και σε όλες τις χώρες. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να αναφέρω και άλλα δύο ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το έργο που κάνουμε στον τα των δικαιώματα. Η αξιοπιστία των βημάτων συζητήσεων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποια είναι η δική μα αξιοπιστία. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να έχουμε ανεξαρτησία, κεραιότητα και αποτελεσματικότητα τη υπηρεσία του ΥΠΑ του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ηνωμένα Έθνη ήταν και παραμένει σημαντικό εταίρο στην θα πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση και διαφάνεια στις διαδικασίες για να διατηρηθεί η αξιοπιστία το ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται για να βοηθήσει την υπηρεσία του είπατε εκπροσώπου για να εκτελέσει τα σημαντικά καθήκοντα. Δηλαδή να εξυπηρετούνται όλοι οι στόχοι της αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες και να δώσουμε τη βοήθεια που χρειάζεται για να εφαρμοστούν οι συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζεται πολιτική υποστήριξη και οικονομική τη αυτή μέσω του Ευρωπαϊκού Εργαλείου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έρθουμε σε εμά του ιδίου. Παγκοσμίω γινόμαστε αντιληπτοί σαν υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαίω καμιά φορά αυτό είναι μια καλή αντίληψη και καλή εικόνα. Κάποιοι άλλοι ε, εταίροι έχουν αμφιβολίε για το ρόλο που παίζουμε, όμω αυτό δεν μα σταματά. Αντιθέτω, αυτό μα δίνει κίνητρο να κινηθούμε περαιτέρω. Ήθελα να πω ότι τελευταία χρόνια τέτοιε αντιλήψει έχουν αμφισβητηθεί η, τα γεγονότα τα πρόσφατα μας θέτουν υποδοκιμασία. Δεν είναι μόνο η κρίση των προσφύγων. Είναι πολλές προκλήσεις πολλών ειδών. Έχουμε και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και το αυξανόμενο συνέστημα της αστάθειας που αισθάνονται οι πολίτες μας. Θα πρέπει να βρουν μια διέξοδο από την κρίση μέσω αλλαγής πολιτικών που θα είναι σημαντική και ορατή. Αυτά Σαφώς δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολη καιρία, αλλά αν λησμονήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρώπης μπορούμε να χάσουμε τα πάντα πριν ακόμα το καταλάβουμε. Εδώ εκπροσωπείται στο ημικύκλιο 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ε, τώρα είσαστε ελάχιστοι βέβαια, αλλά εξακολουθεί να ισχύει. Όλη η πολιτική μας τάξη αντιμετωπίζει σκληρά προβλήματα. Για, οι πολιτικές μας πρέπει να αντικατοπτρίζουν στηρίζουν ότι βέλτιστο διαθέτουμε, ότι βέλτιστο διαθέτει η Ευρώπη και έχουμε επιλογή. Μπορούμε να εστιαστούμε επί των φόβων μας, να τους προωθήσουμε και να τους αφήσουμε να διαλύσουν την Ένωση. Ή μπορούμε να στοιχηματίσουμε στις αξίες που μας ισχυροποίησαν, την ποικιλομορφία μας, τη διαφορά μας, την αλληλεγγύη μας και να ξαναρχίσουμε τους κινητήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι εύκολο σαν έργο, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντέξουμε να, το, να αποτύχουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μογκερίνη. Και τώρα, εξ του ΕΛΚΑ, ο κύριος Ξιμπ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στην σύνταξη αυτού του ψηφίσματος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ θετικό το ότι εφέτος έγκαιρα εγκρίνουμε ένα τέτοιο ψήφισμα προτού ε, θεσπιστούν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής σε σχέση με την θέσπιση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ που υπήρξε αυτή η προθυμία για την ε, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση από πλευρά σας ε, με ανοιχτό τρόπο και για την ε, λήψη υπόψη των σημείων αυτών σε σχέση με την ε, διαβούλευση και με τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά. Μια πολύ σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ένα πολύ μεγάλο κατάλογο προτεραιοτήτων βλέπουμε που είναι τόσο σημαντικά θέματα για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ανήκουν σε αυτά και η λειτουργούσα αυτοδιοίκηση και επίσης η λειτουργία επίσης του Διεθνούς Δικαστηρίου και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και για την καταπολέμηση της θανατικής πηγής ή τουλάχιστον ένα μορατόριο για την μη εκτέλεση θανατικών ποινών. Σεβασμός λοιπόν των δικαιωμάτων του ανθρώπου που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα παγκόσμια. Ας λάβουμε υπόψη επίσης, ας σκεφτούμε και την, προσφυγή, την κρίση με τους πρόσφυγες. Έχουμε πάρα πολλά και συνδέεται και με την ανθρωπιστική κρίση, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε πολλά πολυσχηδή επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι και η ανεξιθρησκεία, η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διασφαλίζεται, διακηρύσσεται αυτή η ελευθερία και τονίζεται η σπουδαιότητά της, η εμβέλειά της πρέπει να πούμε ότι έχουμε ενώπιόν μας την μεγαλύτερη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκόσμιο διεθνούς χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για το ότι τηρήσατε τον χρόνο. Πώς στη συνέχεια έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά και την ύπατη εκπρόσωπο για τα όσα θετικά μας εξέθεσε που καταδεικνύουν τον μεγάλο σεβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου από πλευρά της. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που εκπώνησαν και αυτή την πρόταση ψηφίσματος και που κατέδειξαν με αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντικό είναι αυτό το ψήφισμα και πόσο μεγάλη η εμβέλειά του. Σημαντικό αυτό το θέμα για το να ασχολείται κανείς με τα δικαιώματα του ανθρώπου τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Αυτό το ψήφισμα καταδεικνύει ότι το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη και την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκόσμια και τα θεμελιώδη δικαιώματα βρίσκονται ως ανώτατη προτεραιότητα για την εξωτερική μας πολιτική πάνω πάνω. Υπάρχει δεδομένος λοιπόν ο σεβασμός του Ευρωκοινοβουλίου για αυτά τα δικαιώματα. Σε περιόδους ε, κρίσης καταδεικνύεται ότι δεν επιτρέπεται να αναμένουμε και να καθυστερούμε. Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει δραστήρια να δράσουμε. Είναι το θεμέλιο ακρογωνιαίος λίθος τα δικαιώματα του ανθρώπου για οποιαδήποτε δράση. Αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων των προσφύγων έχει τεράστια σημασία την διασφάλιση διάβλων ή διαδρόμων για την, ε, να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια οι πρόσφυγες είναι ύψης της σημασίας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην υγεία, στην υγειονομική περίθαλψη ως δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να μεριμνήσουμε ότι οι γυναίκες θα είναι ίσες με τους άνδρες. Πρόκειται στο ψήφισμα επίσης και για τα δικαιώματα των παιδιών και για τους κλιματικούς πρόσφυγες και για τους εσωτερικά εκτοπισμένους πολίτες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες παραβιάσεις και παραβάσεις όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Στο ψήφισμα αφορώνται ιδιαίτερα χώρες που παρατηρούνται σε αυτές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πέρα από όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε αυτό το ψήφισμα και έτσι ο έκτακτος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου θα μπορέσει να διαδραματίσει ένα ρόλο ώστε να υπάρξει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την κατάσταση σε σχέση με τα ότι τεκταίνεται στην Παλαιστίνη και να μην παρακολύεται η δράση εκεί των παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε επίσης οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα του ανθρώπου που παγκόσμια δραστηριοποιούν δραστηριοποιούνται ή και στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται άοχνα να ληφθούν υπόψη οι, ε, τα δικά τους συμφέροντα. Να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα όταν θα συνέρθουμε στη Γενέβη ε, προσεχώς ή να αναλάβει τον ρόλο της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος, ως προπομπός. Θα έπρεπε να είμαστε ένας ισχυρός εταίρος στην διεθνή σκηνή παγκόσμια στη συνεργασία υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φων έχει τον λόγο παρακαλώ. Η κυρία Φωνστόρχ, ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητάμε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα Ηνωμένα Έθνη. Και πολλές φορές ε, λέμε ή δρούμε σαν να ήταν ανεξάρτητο κράτος η Ευρωπαϊκή Ένωση με ξεχωριστή εξωτερική πολιτική από πλευρά του. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια. Όμως ε, θα ήθελα να σας καλέσω θερμά για κάποια θέματα όσον αφορά τα θέματα αυτά κυρία Μογκερίνη τους διωγμούς των χριστιανών, την καταδίωξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, να το θέσετε ως ε, ύψης της προτεραιότητας θέμα από πλευρά σας. Η διωγμή των χριστιανών, χριστιανικών πληθυσμών πρέπει να βρίσκεται ως ανώτατο ε, ιεραρχημένο ε, θέμα στις προτεραιότητες που θα έχετε θεσπίσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωνστόρ. Στην συνέχεια θα λάβει τον ε, λόγο συμφωνούμε, είμαστε κάποιοι αρκετοί ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια ακόμα. Η κυρία Μπεατρίς Μπετσέρα Μπάστερετσέα, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Μογγελίνη. Ευχαριστώ για το, τη ε, στεναρότητά σας. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου που προσυπογράφουν αυτό το κοινό ψήφισμα. Ιδιαίτερα από πλευρά συζητού Κρίς ε, για την ε, σαφήνεια όσον αφορά τις κοινέ αξίες. Μόνο έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες να τους εκπροσωπούμε. Σε σχέση με το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστασία των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τα υποψήφια κράτη. Εφόσον έχουν καθοριστεί θα πρέπει να μπορούν επί τρία έτη να παρατηρηθούν. Οποιοςδήποτε ε, πολίτης το ακούσει αυτό και βλέπει ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή η Βενεζουέλα αποτελούν μέρος διαρωτώνται οι πολίτες πώς είναι δυνατόν χώρες που παραβιάζουν συστηματικά τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα να βοηθήσουν για το σεβασμό τους. Θα πρέπει εδώ για την ελευθερία της έκφρασης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή το κράτος δικαίου πώς γίνεται αυτό όταν υπάρχουν δεκάδες κρατούμενοι οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές επειδή διαφωνούν με την κυβέρνηση, διαφωνούσαν με την κυβέρνηση του κυρίου Μαδούρο και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ ρεκόρ εκτελέσεων θανατικών εκτελέσεων θα είχε το ε, θα είχαν το δικαίωμα τα, Ηνωμένα Έθνη να πάψουν, να καταργήσουν την ιδιότητα μελών σε αυτό το ε, όργανο αυτών των κρατών. Όταν πρόκειται για τη Σαουδική Αραβία ή τη Βενεζουέλα για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπονομεύουν την αξιοπιστία αυτών των οργάνων παγκόσμια αυτές οι χώρες. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα ε, και εμείς ε, οι Ευρωπαίοι. Όταν για παράδειγμα δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ της εκλογής χωρών που δεν δεν υλοποιούν τα αναγκαία, τις αναγκαίες απαιτήσεις για να αποτελούν μέρος αυτών των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και στην συνέχεια θα μπορέσει να λάβει τον λόγο εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς η κυρία Βεζά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε για αυτά τα θέματα σε αυτή εδώ το σώμα. Συνήθως ψηφίζουμε ψηφίσματα ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι σύνοδοι του ΟΗΕ χωρίς να λεφθεί υπόψη δική μας σε διάταξη. Αυτή τη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει ένα ψήφισμα νωρίτερα, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες της Επιτροπής του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε ε, έτσι. Δεν σας αμφισβητώ εσάς κυρία Υπατή. Πρόσωπα αντιθέτως επικριτώ την επέμβασή σας. Τα κράτη-μέλη έχουν κάθε κέρδος από το να εξετάζουν προσεκτικά και να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, ιδιαίτερα για την, ε, ε, το χρέη, τα δικαιώματα των γυναικών, την οικονομία κτλ κτλ. Χάνουμε την αξιοπιστία μας όταν δεν μπορούμε και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε από τις τρίτες χώρες να συμμορφώνονται προς δικαιώματα τα οποία οι τα ίδια δεν σέβονται. Ε, για όλους αυτούς τους λόγους η Γκουε αποφάσισε να μην συνδεθεί με αυτό το ψήφισμα και θα τηρήσει αποχή στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων η κυρία Βάρβαρα Λόχμπιλερ. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, το ψήφισμά μας ε, όσον αφορά το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ετοιμάστηκε έγκαιρα και ελπίζω ότι η αντιπροσωπεία μας αυτές τις συστάσεις θα τις λάβει υπόψη στις προτεραιότητές της στις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι το σφαιρικό παγκόσμιο όργανο θεσμικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν ενεργά να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις και στις εργασίες είτε για την κατάσταση επιμέρους χωρών είτε για την εξέλιξη των θεμάτων των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ζητάμε επίση ε, και χρηματοδοτικά να υποστηρίξει το έργο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του με αυτέ τι δράσει. Δυστυχώ σε αυτό τον φορέα, σε αυτό το θεσμικό όργανο συμμετέχουν κυβερνήσει οι οποίε έχουν ολέθριε επιδόσει όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Γι' αυτό θα πρέπει στεναρά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά στην εκλογή και συμμετοχή τέτοιου είδους κρατών σε αυτό το όργανο. Μπορεί να κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλεί με μία φωνή ενωμένα. Ακούμε πολλές φορές τις επικρίσεις ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι εργαλεία ε, υπεριαλιστικής ανάμειξης στα εσωτερικά των κρατών. Γι' αυτό είναι σημαντικό ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει από κοινού κυβερνήσεις να προωθήσει ψηφίσματα, για παράδειγμα ψήφισμα για την ε, ποιότητα του πόσιμου νερού και τι υγειονομικέ ε, υπηρεσίε λυπούμεθα ότι υπάρχει πολλές φορές αρνητική στάση για κάποια θέματα που ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου ε, είναι πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την υπερχρέωση ε, χωρών και την υπερβολική ε, επιβάρυνσή τους των χωρών του Νότου. Είναι πολύ θετικό λοιπόν να τοποθετηθούμε στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ και εγώ πολύ για τις διαβουλεύσεις όπως διεξήχθησαν. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστούμε και στη συνέχεια κοράω παρακαλώ. Έχετε τον Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε. Η σημερινή συζήτηση μας δίνει δυνατότητα να αναφερθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, αλλά είναι κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ευθύνε σαν Ευρωπαίοι. Το ψήφισμα είναι υποστηρίζουμε το, ψήφισμα προς θέλει να προστατεύσουμε τους, τους ταγενείς ε, πληθυσμούς, να απαγωγείται η αρπαγή γεών, το land grabbing και θα πρέπει να ζουν σε κοινωνικέ συνθήκε και οικονομικέ αξιοπρεπεί. Κράζουμε μεγάλη ανησυχία, διότι μέλη του Συμβουλίου πολύ συχνά επιλέγονται μεταξύ χωρών ε, που δεν έχουν, προστατεύουν τα, δικαιώματα, όπω η Ρωσία, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Αιθιοπία. Δεν προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι απειλέ κατά των δικαιωμάτων είναι σε μεγάλη κλίμακα, όχι μόνο τρομοκρατία και των διαφόρων συναφών φαινόμενων όπω ε, θανατικέ εκτελέσει, ε, εκείνο που συνεργάζονται με του ακτιβιστέ, ε, συλλήψει πολιτικών, αντιφρονούντων κλπ. Έχουμε και τι συνέπειε και τη αλλαγή του κλίματο που συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα. Με αυτό το ψήφισμα ζητάμε από το Συμβούλιο τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΟΗΕ να ανταποκρίνεται στο ύψο των καθηκών μα τεθήκαν. Ελπίζουμε το 2016 να είναι πιο θετικό έτος σε σχέση με το 2015. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Άνεμας. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε μια πολύ μεγάλη, γεμάτη και κοπιαστική ημέρα που διανύσαμε μέχρι τώρα τα 700, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέποντας γύρω μου στην αίθουσα πρέπει να πω με τους όσους ε, βλέπω παρόντες ε, μπορούμε παρόλα αυτά να συναγάγουμε πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά δεν θέλω να ακουστώ ή να απηχείτε κινησμός από αυτή μου την παρατήρηση. Δεν πρέπει να υπάρξει λανθασμένη ερμηνεία του Σέγγεν και των δικαιωμάτων των προσφύγων όσον αφορά την ε, σύμβαση της Γενέβης και βλέποντας πόσο έχει η κατάσταση εκφύγει κάθε ελέγχου βλέπουμε στην κολονία με φρικτό τρόπο πως τα δικαιώματα του ανθρώπου ποδοπατήθηκαν και ποδοπατήθηκαν μαζικά από τα όσα συνέβησαν εκεί στην κολονία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπορούν σε ένα σταθές περιβάλλον να ευδοκιμήσουν. Χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον και με ανθρώπους διαφορετικούς από εκείνους που έκαναν τα όσα έκαναν στην κολονία. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Επιτίδιος μεγαλύτερου παίχτε στην παγκόσμια σκακέρα με δυνατότητε που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τι διεθνεί εξελίξει. πρέπει λοιπόν να συνεργάζεται στενά με τον οηε για τον χειρισμό των σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. ένα από αυτά το πιο σοβαρό και επίγον είναι το μεταναστευτικό. για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε με πραγματιστική προσέγγιση. δεν νοείται δηλαδή να προσπαθούμε να φιλοξενήσουμε τους μετανάστες στην ευρώπη και παράλληλα να μην προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις αιτίες που προκαλούν τη μετανάστευση ώστε να τη σταματήσουμε. επίσης δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και να τους επιτρέπουμε να έχουν παραβατική συμπεριφορά στις χώρες στις οποίες φιλοξενούνται. επιπλέον δεν κερδίζουμε κάτι εάν καταδικάζουμε μεν την παράνομη μετακίνηση και διακίνηση των ανθρώπων και αφήνουμε ανεξέλεγκτους να δρουν τους ε, παρανόμους διακινητές τέλος δεν δείχνουμε ούτε σοβαρότητα ούτε αποφασιστικότητα όταν επιτρέπουμε στην τουρκία να περιπέζει την ευρωπαϊκή ένωση ότι δήθεν θέλει να συμβάλει στην επίλυση του μεταναστευτικού και παράλληλα να την ανεχόμαστε να μας εκβιάζει για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της ε, εντάξεώς της. Σας ευχαριστώ στα ελληνικά. Στη συνέχεια ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επενθυμίσω ότι εδώ και ένα μήνα συζητήσαμε και θετήσαμε μεγάλη πλειοψηφία εδώ την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ένωσης επί του θέματος. Έκτοτε και συνεπώς δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί αφιερών, που τόσο σύντομα ψηφίζουμε ένα κείμενο, τόσο σύντομα μετά, που μέχρι κάποιο βαθμό είναι παρόμοιο με την ετήσια έκθεση. Σε αυτό το ψήφισμα, το οποίο θεωρείται ότι εκφράζει τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά τι προτεραιότητε τη Ένωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όλα τα θέματα που έχουν οδήποτε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα καλύπτονται από γυναίκες, ε, ε, αθλητισμό, εμπόριο, μη επανδρομένα οχήματα. Και μέσω του ψηφισματο τελικά παραμορφώνουμε πλήρως ε, το νόημα της έννοιας προτεραιότητα και επαναλαμβάνουμε μια δουλειά που ήδη έχει γίνει. Λοιπόν, είναι ουσιαστικό κατά την άποψή μου τον επόμενο χρόνο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτών των θεμάτων να είναι συντομότερο και να συνάδει με τον στόχο του περισσότερο. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε πέντε προτεραιότητες και να σταματήσουμε εκεί για τις θέσει του Ευρωκοινοβουλίου επί όλων των άλλων θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε την ετήσια έκθεση. Δεύτερο σημείο επί το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό που αφορά το δεύτερο τμήμα του κειμένου που καλύπτει θεωρητικό πώ τον κατάλογο των χωρών υποπεριοδική γενική εξέταση. Διότι εκεί υπάρχει ασυνέπεια προφανέ, κατάφορη κατόπιν επιμονή αριστερά που ήθελε και δεν είναι η πρώτη φορά γι' αυτό να στοχεύσει, να στοχεύσει και να στιγματίσει το Ισραήλ, έχουμε εισαγάγει εντό του καταλάγου ε, την ενευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή. παράγραφος 89, εξυπακούεται ότι δεν είναι μια χώρα και ότι η περιοδική εξέταση η γενική δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αν θέλουμε σαν Ευρωκοινοβούλιο να λαμβανόμαστε σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδου συνέπειε. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα του ΕΛΚ αποφάσισε να διεξαγάγει ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτήν την παράγραφο. Και αν αυτή η παράγραφο δεν διαγραφεί, θα καταψηφίσουμε το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρίτσαρτ Χάουιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν εισηγητή για την εταιρική ευθύνη, προσβλέπω την επόμενη του Συμβουλίου του ΟΗΕ και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου μέσω αντιπροσωπεία και θέλω να προωθήσουμε τι προτεραιότητέ μα. Επιχειρήσει και ανθρώπινα δικαιώματα. Παράγραφο 28 του ψηφίσματο. Λέμε σαφώ, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή θα πρέπει επικοδομητικά να κινηθούν στη διακυβερνητική ομάδα εργασία για ένα μέσο νομικά δεσμευτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προηγουμένω έφευγε από την αίθουσα, μετά την πρώτη μέρα έφυγε. Και αυτό ίσω να επεκρίθη μάλιστα στην έκθεση τη ομάδα εργασία του ΟΗΕ που πρόκειται να παρουσιαστεί τον μήνα Μάρτιο το να αποφύγουμε και να μποϊκοτάρουμε ένα μηχανισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι η θέση της Ευρώπης. Το ψήφισμά μας καθιστά σαφές ότι η συμμετοχή σε μια ανοιχτή ομάδα εργασίας δεν είναι εναλλακτική όσον αφορά τη, λογοδοσία που επιδιώκει ο ύπατος εκπρόσωπος ούτε εναλλακτική στην πρόθεση των αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα κράτη-μέλη εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν ολοκληρώνοντας τα εθνικά σχέδια δράσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να εξετάσει το δεχόμενο ψηφίσματο στη Γενέβη που θα επικρίνει την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ. Αυτό είναι το μονοπάτι της αντιπαράθεσης. Αυτό το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει με κάτι τέτοιο για την ομάδα μου θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ με όλε τι προτάσει που συζητήθηκαν στην ομάδα εργασία. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν για κάθε επιχείρηση και όχι μόνο για την διεθνή συνεργασία και τι διεθνεί επιχειρήσει. Θα πρέπει να είναι στην αίθουσα όμω η Ευρώπη, διπλωματικά να εκφράζει τη διαφωνία τη και να δείχνει στους άλλους η Ευρώπη αυτό που πολύ συχνά τους λέμε να κάνουν. Δηλαδή να είναι έτοιμοι να ακούσουν σε διαφορετικές απόψεις. Και τέλος, Απευθυνόμαστε στον κύριο Μπρέντα που σε την παράγραφο 89. Ε, το κάνει η βασική ψηφοφορία για την ομάδα του και είπε ότι θα καταψηφίσουν το ψήφισμα αν διατηρηθεί αυτή η παράγραφό. Τι λέει η παράγραφος. Υποστηρίζει συμμόρφωση με τη Διεθνή Νόμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ζητά τη βιωσιμότητα τη λύση των δύο κρατών και ζητά υποστήριξη για τον ειδικό εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη εδάφη τη Παλαιστίνη. Και του λέω και σε εκείνο και στην ομάδα του Έχουμε συνένεση να προχωρήσουμε όσον αφορά την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πιστεύουμε ότι η υπερψήφιση των αρχών είναι σωστό για να πετύχουμε ειρήνη μεταξύ ειρήνης και Παλαιστίνης. Αν αυτός και η ομάδα του επιλέξουν να διαφωνήσουν επ' αυτού κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος, τότε εκείνοι σφάλουν. Thank you. Ε, Σας ευχαριστώ. Κυρίες Βάουτμαν, σε παρακαλώ, έχει στη συνέχεια τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βάουτμαν, κυρία Μογκερίνη. Είναι προχωρημένη η ώρα, δυστυχώς δεν παρίστανται πολλοί συνάδελφοι. Κάνουμε όμως λόγο για ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχουμε το θέμα της έγκρισης του ψηφίσματος με το οποίο τοποθετούμεθα επ' αυτών των θεμάτων. Ε, τρεις παρατηρήσεις ως μέλος της ΑΛΤΕ θα ήθελα να γίνει λόγος και για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τις ε, ε, σεξουαλικές επιλογές και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της έκθρωσης μετά από σεξουαλική βία η επίθεση. Γνωρίζω ότι συμμερίζεστε αυτή την ε, άποψη κυρία Μογκερίνη. Δικαιώματα των παιδιών, Save the Children, χιλιάδες, μυριάδες παιδιά οδηγούνται σε αυτούς ε, τους ε, μεταξύ αυτών των προσφύγων. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε να παγώσουν τα παιδιά μέσα στα, στις μάζες των προσφύγων και θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά σήμερα αυτό ακόμα και αν κάποιοι δεν θέλουν να το ακούσουν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη δεν θέλουμε να ε, στιγματίσουμε το Ισραήλ θα ήθελα όμως να αναφερθούμε στα σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με αυτή τη χώρα σας ευχαριστούμε πολύ στη συνέχεια Στυρ έχετε τον λόγο παρακαλώ 1,5 λεπτό ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε θα ήθελα να αναφέρω ότι θα ήταν κρίμα πραγματικά η ομάδα μας να μην μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ψήφισμα λόγω του ότι ε, για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή υπάρχουν κάποιες ε, αναφορές που δεν είναι απόλυτα συμμετρικές. Και στο εδάφιο του ψηφίσματος που αφορά για παράδειγμα τις ε, συνταγματικές ε, αναθεωρήσεις ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην Αφρική για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν ως πρόσχημα χώρες για να αγνοούν τα δικαιώματα πολλές φορές και να ευνοούν κάποιους και αυτό αποτελεί έναυσμα στη βία. Γίνεται λόγος και για τον Μπουρούντι. Δεν είναι όμως το μόνο παράδειγμα. Δυστυχώς υφίσταται μια τάση με αυτή την δραστηριοποίηση, δηλαδή μια οπισθοποίηση στην εξέλιξη αυτών των χωρών. Και αυτό που οδηγεί, οδηγεί στην παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών που κατάφορα παραβιάζονται πολλές φορές τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το κυβερνών κόμμα κερδίζει πάνω, με πάνω από 80% εκλογές για παράδειγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουμε υπόψη τέτοιου είδους ε, δράσεις από πλευράς ε, κομμάτων της Αφρικής, ε, κυβερνητικών κομμάτων και των καταχρήσεών τους. Και η ανάπτυξη όσον αφορά τον στόχο 16 θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ανάπτυξη το 2016 με συγχωρείτε από πλευράς μας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Και στη συνέχεια τώρα θα έχετε τον λόγο παρακαλώ Στυρ. Η ε, κυρία Κινίτσι. I'm Λείπει. Λυπούμε. Η κυρία Τερέζα Κομοντίνη Κάκια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να στρέψουμε με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματά τους. Θα πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή, ε, το, η υλοποίηση των δικαιωμάτων χωλαίνει πολλές φορές. Βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό το οποίο θα έπρεπε πάντα στις κοινωνίες μας. Είναι όμως πλήρη μέλη των κοινωνιών μας. Ο ευάλωτος χαρακτήρας τους όμως ε, τα καθιστά θύματα σε σχέση με ε, τον περίγυρό του. Πρέπει η ε, αρνητική μεταχείριση, η εκμετάλλευση να αποφεύγεται. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσει το έργο της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι μόνο μια πολλές, ε, ε, η πιο επικυρωμένη από τους περισσότερους σύμβαση, αλλά η σύμβαση εκείνη η οποία θα εφαρμοστεί κιόλα από όλους. Επίσης, οδεύοντας προς ένα καλύτερο μέλλον, αυτά τα παιδιά με μεταξύ των ε, προσφύγων υφίστανται τα πάνδυνα και θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Είναι καθήκον μας να, να καταπολεμήσουμε την ομότητα εις βάρος αυτών των παιδιών. Πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ και στη συνέχεια η κυρία Χιμένεθ Μπεθερή Μπάριο ε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα πρέπει να δράσουμε για να υπερασπιστούμε εκείνους ε, που πάσχουν, ε, που υφίστανται διώξεις και στέρηση της ελευθερίας τους. Επίσης για τόσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα παρότι το Κοινοβούλιο σχέση με την αποστολή σε αυτή τη χώρα <clears throat> το έλκα σε σχέση με την ε, δράση μας για την ε, Βενεζουέλα σε αυτή την ιστορική στιγμή εκείνων που ε, ήταν υπέρ της ελευθερίας που κατάφεραν να κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση έναντι εκείνων που ήταν κατά της ελευθερίας όλα αυτά όμως χάνουν την αξία τους όταν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αγνοεί τα δικαιώματα αυτά και την αμνηστία που απαιτεί την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται στις φυλακές από την κυβέρνηση της Βενεζουέλα. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο να πιέσουν τις αρχές της Βενεζουέλας για την απελευθέρωση των φυλακισμένων. Και ο Μαζούρο, Μαδούρο συνεχίζει χωρίς να ακούει τις κραυγές των πολιτών του που απαιτούν την ελευθερία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Κούκαν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί είπατε εκπρόσωπε. Φέτος έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη η ίδια αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου προβλήματα όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία και η αυξανόμενη αστάθεια στη γειτονιά μας. Γι' αυτό το λόγο τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι πιο επίγοντα ακόμα και θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες για το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η βάση της σύγχρονης Ευρώπης και θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα αυτό στον ΟΗΕ, να ηγηθούμε μάλιστα. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο θεματολόγιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τη μετανάστευση θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια και να συμβάλλουμε στην μείωση της φτώχειας σε κρίσιμες περιοχές του κόσμου. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα όσον αφορά την καταπολέμηση των δικτύων διακινήσεως ανθρώπων και να ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βίντα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία, είπατε πρόσωπε για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εντολή της κοινότητας των εθνών για να, δράσει, να δράσουν και θα πρέπει και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λυπούμαστε που δεν έχει ρυθμιστεί με τον καλύτερο τρόπο η ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να μεριμνήσουμε και να δράσουμε ώστε να μπορέσουν και οι εκπρόσωποι των πολιτών ε, να εμπλέκονται και να συμμετάσχουν. Σημαντικό θα ήταν να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και στο κρατικό εθνικό επίπεδο αλλά και στο περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης και από πλευράς ε, των κύκλων της οικονομίας να είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δυστυχώς όμως ε, παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και ατιμόρυτα οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πολιεθνικές διεθνικέ περιφρονούν τα δικαιώματα του ανθρώπου ενώ θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πάντα σεβαστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νότης Μαριάς παρακαλώ έχει τον λόγο. Πρόεδρε, στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιληφθούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία αλλά και στα Σκόπια. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε δάτρω με της ευκαιρίας να τονίσω την πλήρη και κάθετη αντίθεσή μου με την πρωτοβουλία της ευρωβουλευτού από την κροατία marianas petir να προχωρήσει στη δημιουργία ανεπίσημης ομάδας φιλίας με το όνομα φίλοι της μακεδονίας με στόχο τη στήριξη των σκοπίων. υπενθυμίζουμε στην εν λόγω ευρωβουλευτή ότι τα σκόπια αναγνωρίζονται από την ευρωπαϊκή ένωση με την προσωρινή ονομασία ΦΥΡΟΜ και με κανένα άλλο όνομα. να γνωρίζει εν λόγω ευρωβουλευτής ότι δεν θα επιτρέψουμε στα σκόπια και τους κάθε λογής συνοδοιπόρους του να οικειοποιηθούν το όνομα της μακεδονίας μας. καταγγέλλω λοιπόν ενώπιον του σώματος την προκλητική και συνάμα παράνομη δημιουργία της φιλοσκοπιανής ομάδας με τον τίτλο φίλοι της μακεδονίας και ζητώ από τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου μάρτιν σούλτς να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή και στην εν λόγω υπόθεση των αποφάσεων του οηε που σχετίζονται με την ονομασία των σκοπίων. Ευχαριστώ. παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρία, γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια άτυπη ομάδα και η οποία υπήρχε και κατά το παρελθόν. Δεν είναι τίποτα καινούριο η ύπαρξή τη. Αυτό αφενό. Αφετέρου, δεν έχει καμιά σχέση με το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα, εντάξει. Πολύ σύντομα παρακαλώ εσείς κύριε Μαρία. Να απευθυνθώ στον συνάδελφο και να του πω ότι έθεσα ένα σοβαρό θέμα. Τα Σκόπια αναγνωρίζονται με το όνομα φύρομ εσείς παρανόμως χρησιμοποιείτε το όνομα μακεδονία και αυτό που κάνετε όσοι κάνετε αυτή την ομάδα να γνωρίζετε ότι είναι παραβίαση και του τρόπου λειτουργίας της ευρωπαϊκής ένωσης που αναγνωρίζει τα σκόπια με το όνομα φύρομ. να το καταλάβετε αυτό μια για πάντα. Ε, και τώρα κυρία Μογκερίνη, είπατε εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Δεν θα μακρηγορήσω ώστε να μην μείνουμε για πολύ ακόμα σε το τιμικύκλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα όσους έμειναν στο θέμα της ε, συζήτησης. Ναι. Και που επένεσαν την Κομισιόν για το έργο μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. πολύ, από σας είπαν ότι ε, είναι μια αρχή να προστατεύουμε και να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ένωσης. Και σε αυτό το έργο θα πρέπει να σας πω ότι η υποστήριξη αλλά και η κατεύθυνση, η καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να χρησιμοποιήσουμε την τα... τα μέσα ε, εξωτερικής δράσης ε, από κοινού ώστε να συμπληρώσουμε και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας με κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου. Κάποιες φορές αυτό είναι προφανές, κάποιες φορές λιγότερο προφανές, πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις είτε είναι μεμονωμένοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μεγάλες υποθέσεις οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι μακρύς ο κατάλογος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει τη διαφορά όταν με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, ε, συνεργαζόμαστε. Η κατάσταση είναι δύσκολη ε, αλλά υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αμέσω συμφέροντά μα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα για σταθερότητα εάν δεν υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαφώ και φέρουμε ευθύνη εντό των συνόρων μα αλλά και εκτό. Και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη στήριξη του και προσωπικά να ευχαριστήσω και τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη, τον ε, εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε να προωθήσουμε από κοινού αυτή ε, την υπόθεση. Σας εύχομαι καλό, καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε.